Okay, Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Καλώς ορίσατε και πάλι στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, να σας πω ότι δεν ήμουν εδώ στην αρχή της χθεσινής μας συνεδρίασης γιατί είχε καθυστέρηση το Eurostar και γι' αυτό καθυστέρησα να έρθω. Σίγουρα όμως όλοι χαρήκατε όταν μάθατε, όπως και εγώ χάρηκα, όταν μάθατε ότι οι δύο από τις υποψηφιότητε για τα βραβεία Ζαχάροφ, ο δόκτωρ Ντένις Μακουέκη και η Νάντια Μουράτ, είναι αυτοί στους οποίους απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. Εξαιρετικά νέα για την δουλειά της Επιτροπής μας, η οποία αναδεικνύει αναπτυξιακά ζητήματα και εργάζεται για να δοθεί ένα τέρμα, ένα τέλος στη βία εναντίον των γυναικών. Αυτά λοιπόν ήταν τα καλά νέα της περασμένης εβδομάδας, το τέλος της περασμένης εβδομάδας. Καλούμαστε όμως τώρα να ξεκινήσουμε τη δουλειά και δει την ψηφοφορία. Και τώρα ε, βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης ψηφιοποίηση για την μείωση της φτώχειας μέσω της τεχνολογίας. Θα ψηφίσουμε και εντός ολίγου θα δώσω το λόγο στον εισηγητή Βέντερ πριν το ξεκινήσουμε όμως να ε, κάνουμε ένα τεστ των μηχανημάτων, να δούμε αν δουλεύουν, παρακαλώ να πατήσετε τα κουμπιά για να ελέγξουμε ότι λειτουργεί σωστά το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας. 18 έχουν τοποθετήσει τις κάρτες τους, δεν είναι και πολλοί. Στην Επιτροπή μας, σύμφωνα με το μηχάνημα, 15 ψήφισαν, τώρα 20 έβαλαν την κάρτα τους, 17 ψήφισαν. Ποιος δεν ψήφισε, Παρακαλώ βάλτε τις κάρτες και ψηφίστε υπέρ σε αυτή την ε, δοκιμαστική ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία απλά να ελέγξει ο καθένας ότι το μηχάνημά του δουλεύει. Να μην υπάρχει κάποιος που να έχει βάλει την κάρτα του και να μην έχει ψηφίσει, να μην έχει πατήσει το κουμπί. Για να δούμε ότι όλα τα μηχανήματα δουλεύουν. Άρα 22 ψήφοι, όλα τα μηχανήματα δουλεύουν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δοκιμαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όπως έλεγα λοιπόν, είμαστε στο σημείο 15 τη ημερήσιας διάταξης, ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη, μείωση της φτώχειας μέσα από την τεχνολογία. Μπόγκταν, μήπως θα θέλατε να πάρετε το λόγο. Όχι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. hang on. Okay, I think all Νομίζω ότι όλα τα μηχανήματα λειτουργούν για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το ΕΛΚ έχει 8 ψήφου. Okay. Μπόγκταν, δεν θέλετε κάτι να πείτε. Όχι. Καλώς. Ξέρω ότι είχε γίνει πολύ σκληρή δουλειά για να καταλήξουμε στην έκθεση αυτή και έχετε, βρεθεί, έχετε καταλήξει σε πολλές συμβαστικές τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ της πρώτης συμβαστικής υποτροπολογίας. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την συμβιβαστική 6α, την 6α τροπολογία για τη νέα διατύπωση. Νομίζω την έχετε λάβει όλοι, την 6α. Ποιοι είναι υπέρ της 6α. Κατά. Αποχές α, α απορρίπτεται η διατύπωση της 6α. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καλώς. Συμβιβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Όχι, συγγνώμη. 58, έκανα λάθο. Ψηφίσουμε ξεχωριστά την 58, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 58. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 μαζί με την συμβιβαστική 9. Ποιος είναι υπέρ και των δύο. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 11. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 97 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Ε, ηλεκτρονικά, όχι καταπίπτει, συγγνώμη, καταπίπτει. Θα έπρεπε να είχε καταπέσει, δεν την ψηφίζουμε. Πάμε στην 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 99. Η Τερέζα με μπέρδεψε. Είστε υπέρ εσείς. Γι' αυτό έγινε αυτό το προηγούμενο. Πέρα τη ψηφοφορία και ήταν και με μεγάλη πλειοψηφία. 100. Ψηφίζουμε την 100. Υπέρ. Κατά θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 100. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυτά εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά αυτή τη φορά. Πέρασε. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε. Ψηφίζουμε την 112 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 13 ψήφοι υπέρ, 12 κατά. 114 ψηφίζουμε. Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά επαληθεύουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 115 ψηφίσατε όλοι πέρασα εγκρίνεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 119 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, θα το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε την 110, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία, 110 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 132 υπέρ 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε τώρα ε, στους ψήφους της αιτιολογικές αναφορές. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στις ε, αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία υπαριθμών 3 για την αιτιολογική σκέψη Α. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά να το ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε την 5, ελέγχουμε την 5 για την αιτιολογική σκέψη Γ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία υπαριθμών 10. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, ε, ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 11. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Να ελέγξουμε τη 12. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 12. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Με συχνή πλειοψηφία. Η 12 εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε τη 14. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 14. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Ε, επαληθεύουμε την 21. Παρακαλώ, άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Ελέγχουμε την 22, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 22. Ξεκινάμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 24. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά δεν το ξέρω. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συνάδελφοι, να επιστρέψουμε γιατί δεν ψηφίσαμε την 9, την τροπολογία 9. Παρακαλώ να τη βρείτε στα χαρτιά σας. Δεν ξέρω αν, την, ε, αν βρήκαν υπεύθυνοι από κάθε πολιτική ομάδα σε ποια σελίδα βρίσκεται. Βρίσκεται στη σελίδα 8. Τροπολογία Κούλογλου και Λόλα Σάντσεθ. Ε, Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία παριθμών 9. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 9. Που βρίσκεται στη σελίδα 8. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Επιστρέφουμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ονομαστικής ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Βέντε. 19 ε, υπέρ, ένας κατά, 5 αποχές. Μπόγκταν, παρακαλώ. Συγγνώμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά ε, τα στελέχη της Γραμματείας και τους λοιπούς συνεργάτες γιατί κατάφεραν να επιλύσουν πολύ περίπλοκα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη σκληρή τους δουλειά και τους συμβιβασμούς τους. Επόμενο θέμα, το σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης, αναπτυξιακή βοήθεια στο πεδίο της εκπαίδευσης και της παιδείας. Πολύ, σημαντικό γιατί το έδαφος είναι αρκετά ολισθηρό. Ο Βανσάν Πεγιάν είναι ο εισηγητής. Θέλεις κάτι να πεις πριν από την ψηφοφορία. Θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, ευχαριστώ σύντομα και εγώ να ευχαριστήσω τους αδελφούς με τους οποίους συνεργάστηκα με τρόπο συλλογικό για την έκθεση και είμαι πλήρως ικανοποιημένος να ευχαριστήσω και τη γραμματεία της Επιτροπής μας αλλά και των διαφόρων άλλων ομάδων με τις οποίες συνεργαστικά. Όπως και το σύνολο των συναδέλφων να ευχαριστήσω. Ελπίζω η έκθεση αυτή να είναι χρήσιμη επειδή έχουμε μείωση των κονδυλίων και όχι επαρκή προγραμματισμό Έχουμε απώλειες λοιπόν, οπότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, βασική εκπαίδευση η οποία δεν έχει μπει σε αυτή τη μεγάλη αγορά της εκπαίδευσης που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ελπίζω λοιπόν ότι μέχρι το τέλος θα είμαστε θέσει να βοηθήσουμε πολύ κόσμο, τους νέους, τις ΜΚΟ, ε, τα κράτη, κομισιόν, ώστε να αντιμετωπίσουμε μαζί το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχουμε αρκετή δουλειά και με τις συμβαστικές. Ξεκινάμε τη συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26. Τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 και 49 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται να λέξουμε για τις 48 και τις 49 ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τις 48 και τις 49 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 18-7 εγκρίνονται 51-52 ταυτόσημες οι επόμενες υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 51-52 άρχεται νομίζω έχει περάσει αλλά καλού κακού πέρας 18-7 και πάλι πέρασαν Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 κατά πίπτη. Οπότε πάμε στη συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 97 ναι, τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε 109 ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται 109. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται 15-10. 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. και 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Όχι. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Να αλλάξουμε την 9. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ξεκάθαρα. Λέει πρόεδρο, πέρα πέρα, 23 ψήφου με 2. 10 υπέρ κατά απόχέ απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 Την 22 την κάναμε, τη συμβαστική, την ψηφίσαμε. Ναι, ναι, πέρασε. Ε, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η συμβαστική 22. Πάμε τώρα στην τροπολογία 14. 14 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 18 τροπολογία υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογικές αναφορές 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο ονομαστικά όπως έχει τροποποιηθεί. Πέρας. Εγκρίνεται 25 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια Βανσά, πολύ χρήσιμη έκθεση για τις συζητήσεις που θα έχουμε σχετικά με την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο για το Ποιος θα έχουμε βέβαια και τα χρήματα, τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Ωραία. 17. ΠΟΕ. Η συγγύτρια είναι η Λόλα Σάντσες. Θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία τότε. Ξεκινάμε με την τροπολογία 1. Υπέρ. Α, α, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 1. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 δεν ψηφίζουμε. Τροπολογία 14. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται με 15 προς 10. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 15 προς 11. Θα πρέπει να ψηφίσουμε και για την τελευταία πρόταση της α, τροπολογίας 16. Εγκρίνεται. Και προχωράμε τώρα στην 26. Υπέρ, κατά, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έχω την εντύπωση ότι εγκρίνεται. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία υπαριθμό 26. Πέρα τη τροπολογία εγκρίνεται με 16 προς 10. Τροπολογία 27. Υπέρ, κατά. Να ψηφίσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έχουν ψηφίσει όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται με 17 προς 9. Τροπολογία 29. Υπέρ, κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 16 προς 9. Τροπολογία 30. Υπέρ, κατά. Και πάλι να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες, Εγκρίνεται με 16 προς 10. Τροπολογία 31. Υπέρ, κατά, αποχές και πάλι έχουμε πλειοψηφία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Πρέπει τώρα να ψηφίσουμε την τελευταία παράγραφο, πρόταση της ε, τροπολογίας 34 απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 41, άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη ψηφοφορία. Τροπολογία 42. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχω την εντύπωση ότι εγκρίνεται. Ναι, εγκρίνεται με 16 προς 10. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και για τη συμβιβαστική 4. Έχω την εντύπωση ότι εγκρίνεται πέρα στις ψηφοφορίες. Ναι, εγκρίνεται με 15 προς 11. Τροπολογία 55. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58. Υπέρ κατά αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία υπαριθμών 58. Έχω την εντύπωση ότι απορρίπτεται πέρα της ψηφοφορίας. Ναι, απορρίπτεται με 17 προς 9. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα ονομαστικά για τη γνωμοδότηση στο σύνολό τη. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 14 υπέρ, 2 κατά και 10 αποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λόλα Σάντσες. Τελείωσε και αυτή η ψηφοφορία. Έχουμε άλλη μία ψηφοφορία ή αναφορά για την η ενδιάμεση έκθεση είναι το σημείο 18 για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-27. Ναι, είναι η γνωμοδότησή μας προς την Επιτροπή Budget. Η Αριάννα Ζεύκα είναι η η συγγήτρια, θέλετε να πάρετε το λόγο, Αριάννα. Όχι, περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ κατά να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ, για την τροπολογία 10. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται με 16 προς 10. Δεν υπήρχαν αποχές. Για την τροπολογία 3 έχω την εντύπωση ότι εγκρίθηκε. Με συγχωρείτε λέει η πρόεδρος. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 3. Παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με 21 προς 5. Δεν υπάρχουν αποχές. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Η 3. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Έχω την εντύπωση ότι εγκρίνεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ναι, εγκρίνεται με 19 προς 7. Τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ναι, απορρίπτεται. 6 υπέρ 13 κατά. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 13 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 16 προς 10 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 απορρίπτεται Τροπολογία 22. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τροπολογία 23. Υπέρ, κατά, αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται με 16 προς 9. 24 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έχω την αίσθηση ότι εγκρίνεται. πέρα τη ψηφοφορίας εγκρίνεται με 15 προς 10. Τροπολογία 25. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και για την 25. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 25. Πέρας της ψηφοφορίας. Είχατε δίκιο. Ήταν 13 κατά. Είχατε δίκιο που ζητήσατε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 38 υπέρ, κατά, αποχές. Μπορούμε να ψηφίσουμε για την 38 παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. 15 προς 9. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία υπαριθμών 39. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορία. εγκρίνεται με 13 προς 12. Τροπολογία 40 υπέρ κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται με 15 προς 10. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 41 παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες, ναι, εγκρίνεται με 15 προς 10. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 44 και 45, 46 ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 48 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Εγκρίνεται. 51. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τροπολογία 51, παρακαλώ. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 15 προς 10. Τροπολογία 52. Εγκρίνεται. 53 εγκρίνεται. 54 εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε στην ε, γνωμοδότηση, ονοματική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 21 υπέρ 1 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια στην Αριάννα για τη δουλειά της αναλύουμε τώρα τι ψηφίσατε, γιατί θα συζητήσουμε για το πολιετές ε, ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. That concludes the votes, colleagues. Και έτσι ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες. Όσοι φεύγουν παρακαλώ να το πράξουν ησύχως. Συνάδελφοι, προχωρούμε στο σημείο 19 και στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης. Συμφωνία συνεργασίας, εταιρικής σχέσης και ανάπτυξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν. Εκφράζουμε γνωμοδότηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συντάκτης της γνωμοδότηση του κ. Σέγγελ είναι μια συνενετική διαδικασία με συνοδευτικό ψήφισμα για το CAPD για τη συμφωνία αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφγανιστάν και για την έκθεση της κυρίας Φώτιγκα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην ΑΦΕΤ. Η Συμφωνία Συνεργασίας με το Αφγανιστάν υπογράφτηκε το Φεβρουάριο του 2017 και από 1η Δεκεμβρίου εφαρμόζεται προσωρινά. Από την 1η Δεκεμβρίου του 2017. Παρά το γεγονός ότι η Συμφωνία Συνεργασίας έχει στοιχεία που αποτελούν μέρος της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δώσει τη συγκατάθεσή του τόσο αργά όσο ο Φεβρουάριος του 2018. Περιλαμβάνονται και διατάξεις ε, συνεργασία που απαιτούν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Το Αφγανιστάν είναι ένας από τους μεγαλύτερους αποδέκτες αναπτυξιακής βοήθειας και ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτέλεσε το επίκεντρο πολλών συζητήσεων στην Επιτροπή μας. Επομένως, αν θυμάστε καλά, συζητήσαμε για τη διάσκεψη Βρυξελών-Αφγανιστάν το 2016 και την ε, διακήρυξη, την κοινή διακήρυξη για τη μετανάστευση που υπογράφηκε την ίδια μέρη. Διάφορα θέματα συζητήθηκαν και στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου με μέλη της Επιτροπής μας. Θα δώσω το λόγο τώρα στο Φρανκ Έγγελ, ο οποίος ε, είναι πολύ πιο καλά καταρτισμένος από ότι εγώ και μπορεί να μας ενημερώσει ε, για τα δεκτενόμενα. Φρανκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Λίντα. Δεν έχω κάτοψη πιο εμπεριστατωμένη της κατάστασης από ότι εσείς. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Αφγανιστάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτελεί μέρος των σημείων στα οποία είμαστε προσιλωμένοι και θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις περιοχές. Αυτό από τη μία και από την άλλη φαίνεται να μην αλλάζει τίποτα. Και αν τελικά αλλάζει, αλλάζει προς την εσφαλμένη κατεύθυνση. Στην πρώτη παράγραφο λοιπόν της πρότασής μου ε, της πρότασης γνωμοδότησης γράφω αυτό που απεικονίζει σε μεγάλο βαθμό αυτά που δεν δουλεύουν. Από το 2002 μέχρι το 2016 έχουμε δώσει 3,2 ε, βοήθεια. Και παρά τη διεθνή βοήθεια, η οποία δεν είναι καθόλου μελιτέα για μια χώρα που δεν είναι και τεράστια, από το 38% πήγαν 55% των Αφγανών ε, πιο χαμηλά από το κατόφλι της φτώχειας. Όχι μόνο λοιπόν ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, 38% τότε, 55% τώρα, αλλά ε, ζουν και σε όλο μεγαλύτερη ανασφάλεια. Ε, γίνεται προετοιμασία για περιφερειακές εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο φέτος. Την πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά από το 2010 που θα προσέλθουν οι Αφγανοί στις κάλπες για να εκλέξουν μέλη στο κοινοβούλιο τους και περιμένουμε το 1 τρίτο των εκλογικών κέντρων να μην ανοίξουν λόγω της ανασφάλειας που επικρατεί κυρίως το ΒΑΡΑ λόγω της δράσης των Ταλιμπάν και του Ταρεξαμίκ Αυτά μας λέει ο επικεφαλής της αποστολής της αντιπροσωπείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Ο απολογισμός για τα θέματα ασφάλειας των τελευταίων μηνών είναι καταστροφικός. Είναι ο πιο δυσίωνος ε, απολογισμός, 100.000 θύματα, πολίτες, ...1.700 έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα χρόνο Γενικά είναι πολύ δραματική η κατάσταση και μπροστά μας έχουμε το σχέδιο μία συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ημών και του Αφγανιστάν σε θέματα ανάπτυξης. Δεν βλέπω πώς θα αρνεί το μια επιτροπή για την αναπτυξιακή βοήθεια να εγκρίνει μια τέτοια πρωτοβουλία. Λυπούμαστε γιατί δεν ζήτησαν τη γνώμη μας από πριν, πριν τη διατύπωση της πρότασης αυτής συνεργασίας και συμφωνίας συνεργασίας. Έπρεπε να είχαν ζητήσει τη γνώμη μας εκ των προτέρων, έπρεπε να μας είχαν εμπλέξει αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πολλά να συμβάλλουμε και πολλά να συνεισφέρουμε. Πίστευω ακραδάντως ότι είναι καθήκον και υποχρέωσή μας να πούμε ότι πρέπει κανείς να συνεχίσει να στέκεται, να παραστέκεται στο Αφγανιστάν, να στέκεται πλάι στη χώρα αυτή και να προσπαθεί να δρά προς όφελες της χώρας αυτής σε ένα πλαίσιο στο οποίο αυτοί που κυβερνούν και αυτοί που θέλουν να κυβερνούν στη χώρα αυτή το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα δικά τους πλεονεκτήματα και ωφέλη. Κάτι το οποίο δυστυχώς είναι προβληματικό ε, για να, ε, και μας δυσκολεύει, δεν μπορούμε έτσι να αποκτήσουμε εταίρους σε αυτή τη χώρα και να τους αξιοποιήσουμε για να μεταφέρουμε, να λειτουργήσουν αυτοί ως κοιτάλοι και να φτάσει η βοήθειά μας αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτά έχω να πω κατά βάση και γι' αυτό είναι γλυκόπικρα τα συναισθήματα που δημιουργούνται από αυτή τη συμφωνία συνεργασίας, την οποία βεβαίως στηρίζουμε όπως καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ, ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να προσθέσω δύο λόγια στα λόγια του Φρανκ. Είπε ότι η Επιτροπή για την Αναπτυξιακή Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άργησε να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Ίσως με το εργαλείο που συζητήσαμε σήμερα το πρωί στην Ακρόαση θα καταφέρουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία. Αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση. Και εκφράζω και τον Φραντσουλίκα, ο οποίος δεν μπόρεσε τον κύριο Φρουτσούλητσα που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα και ο οποίος είναι σκιώδης εισηγητής για τα θέματα αυτά. Το Αφγανιστάν, λοιπόν, διαβάζω τα λόγια του, αποτελεί χώρα προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Η βία και οι συγκρούσεις έχουν επικυριαρχήσει στη χώρα αυτή και έχουν επηρεάσει την καθημερινότητα και τις ζωές πάρα πολλών Αφγανών πολιτών. Έχουν υπονομεύσει και επιδεινώσει το βιωτικό επίπεδο, έχουν ενισχύσει την πολιτική αστάθεια και ανασφάλεια και έχουν υψώσει εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδι προς την ευημερία ενός πραγματικά εύθραυστου, ευάλωτου κράτους. Πρέπει ε, να αποκαταστήσουμε τις αφές οι προτεραιότητες που είναι οι βασικές κρατικές υπηρεσίες. Ε, στηρίζουμε τον προϋπολογισμό που έχει ως στόχο να αυξήσει τους πόρους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη και στη μείωση της φτώχειας. Στηρίζουμε την καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού μέσω της κρατικής αυτής υπηρεσίας που έχει συσταθεί, της εταιρεία κρατικής, η οποία στοχεύει και στη μείωση της διαφθοράς. Όμως πρέπει να βρεθούν οι σωστές προϋποθέσεις. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα αυτά με θετικό τρόπο έτσι ώστε να επέλθουν θετικές εξελίξεις στη χώρα αυτή. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι λυπούμαστε για την απουσία εποπτείας στοιχειώδους εποπτείας και δημοκρατικού ελέγχου για την ολοκλήρωση των συζητήσεων για τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Και η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αφγανιστάν δεν θα πρέπει να ε, τη βλέπει κανείς μέσα από το πρίσμα της μετανάστευσης και δεν θα πρέπει να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις στη διαχείριση της μετανάστευσης για να έχει συμφωνία συνεργασίας ως Ευρωπαϊκή Ένωση με το Αφγανιστάν η βοήθεια που δίνουμε στη χώρα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι συμβάλλει ε, στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων, καθώς οι γυναίκες ε, συνεχίζουν να προσκρούν σε πολλαπλά εμπόδια που τις παρακολούν και τις εμποδίζουν να έχουν πλήρη συμμετοχή ε, στο γίγνεσθε, το κοινό και το δημόσιο γίγνεσθε αντιμετωπίζουν το κίνδυνο συγκρούσεων και καθημερινής βίας. Σε όλα αυτά τα πεδία πρέπει να σημειωθεί επαρκής πρόοδος και θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην προστασία των γυναικών και στην άσκηση περισσότερων εξουσιών από την πλευρά τους. Και αυτό θα πρέπει να διέπει την καθημερινότητα των σχέσεών μας με το Αφγανιστάν. Ευχαριστώ, η Πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστώ και εγώ. Δεν βλέπω κανείς να ζητά το λόγο. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει το λόγο στη συνέχεια. Έχω εγώ να πω το εξή και να ρωτήσω το εξή. Εμείς είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές. Ποιοι άλλοι είναι δωρητές, ποιοι βοηθούν από τη διεθνή κοινότητα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε φαντάζομαι ότι δίνουν χρήματα, έτσι δεν είναι, και ποια είναι η στρατηγική μας θέση σε σχέση αναλογικά με τους λοιπούς δωρητές. Συμφωνώ με τον Φρανκ και με τον Νόρμπερτ. Πρέπει να ασχοληθούμε πιο ενεργά με τη χώρα αυτή, όμως η πολιτική κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Το επόμενο ερώτημα που έχω να απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εξή. Ποιε είναι οι προοπτικέ τη ειρήνη και τη τελική έκβαση τη αναπτυξιακή βοήθεια, Γιατί πολύ συχνά κάνουμε ένα βήμα μπρο και μετά κάνουμε μισό ή ένα βήμα πίσω. Ε, Ποιε είναι οι προοπτικέ, ε, πώ προβλέπετε τα μελούμενα. Ο Στίβεν Λοκ από την ΤΕΦΚΟ, την Υπηρεσία τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Αλίνα Παππού. Ίσως δεν προφέρω σωστά το όνομά σα και ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω ποιο θέλει πρώτα το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εσείς από πού είστε, η Αλίνα είστε. Από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο εκ μέρους ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη θετική γνωμοδότηση που μας δίνεται για αυτή τη ε, Συμφωνία Συνεργασίας, εταιρική Σχέσης και Ανάπτυξης. Είναι το πρώτο νομικό δεσμευτικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφγανιστάν. Είναι ένα εφαλτήριο, ένα σημείο καμπής, έτσι ώστε οι σχέσεις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή να πάνε σε ένα ανώτερο επίπεδο, ένα σημείο καμπής έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα στη στρατηγική μας στο Αφγανιστάν. Και θα ήθελα να τονίσω ότι η συμφωνία αυτή θα κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει και να ενισχύσει τη μακρό η δέσμευση που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι του λαού του Αφγανιστάν. Θα συμβάλλει στην ειρήνη και στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη. Ένα ειρηνικό και αναπτυσσόμενο Αφγανιστάν είναι κάτι το σημαντικό και για την ευρύτερη περιφέρεια και περιοχή. Εξού και στα τέλη του 2017 υιοθετήσαμε τη νέα στρατηγική για τη χώρα αυτή και τώρα είμαστε σε φάση υλοποίηση και εφαρμογή τη. Η Συμφωνία Συνεργασία λοιπόν, η CIPD, συμβάλλει τα μάλα στην εφαρμογή εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής και της βοήθειας που δίνουμε. Είχαμε προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Συνεργασίας, δύο συναντήσεις φέτος και συζητήσαμε εκεί πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η, η, η ανάληψη περισσότερων εξουσιών από τις γυναίκες. Συζητήσαμε την ισότητα των φύλων, τη συνεργασία, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την περιφερειακή συνεργασία. Ε, περιμένουμε με ανυπομονησία να κυρώσουν τη συμφωνία όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αρχίσουμε να εφαρμόσουμε όλα τα κεφάλαια αυτής και σε όλα τα σχετικά πεδία. Να υπογραμμίσω ότι συμφωνούμε με τους προλαλήσαντες, πράγματι Δυστυχώς το Αφγανιστάν αντιμετωπίζει, συνεχίζει να αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, της οικονομίας, της πολιτικής αρένας, επίκυνται εκλογές, πλησιάζουν οι εκλογές. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχουμε μια ειρηνευτική διαδικασία συμφιλίωσης και επικεφαλής της οποίας θα είναι οι ίδιοι οι Αφγανοί, ο αφγανικός λαός. Και εκφράσαμε την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πλαισιώσει μια πρωτότυπη, μια αυθεντική ειρηνευτική διαδικασία στο Αφγανιστάν με πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Περιμένουμε την ε, Υπουργική Διάσκεψη της Γενέβης για το Αφγανιστάν στα τέλη Νοεμβρίου, το Νοέμβριο. Είναι η επόμενη μετά τη διάσκεψη των Βρυξελών για το, Βρυξελ, για το Αφγανιστάν που έλαβε χώρα το 2016. Στη Γενέβη λοιπόν θα κάνουμε αποτίμηση της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα αυτή από τη διάσκεψη των Βρυξελών μέχρι και σήμερα, δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια. Και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια περιφερειακή συνένεση για ε, περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Από την πλευρά μας δηλαδή κάνουμε ό,τι μπορούμε και βεβαίως θα τηρούμε ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τέσσερις γρήγορες παρατηρήσεις από εμά αν επιτρέπετε. Υπόθηκε ότι είχαμε μια αύξηση του επίπεδου της στόχιας στο Αφγανιστάν. Είναι σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση. Αφενός βλέπουμε μια ξεκάθαρη πρόοδο όσον αφορά τους κοινωνικούς δείκτες, δηλαδή δείκτες αλφαβητισμού, θυσιμότητα βρεφών και ε, μητέρων δράση κυβέρνησης, εταιρικέ σχέσεις, όλα αυτά βέβαια συνοδεύονται από την ανασφάλεια, τη διατροφική και την αύξηση της φτώχειας, κατά το οποίο εξηγεί βεβαίως και την κακή κατάσταση της οικονομίας. Έχουμε υποβάθμιση της ε, ασφάλειας, εκτοπισμούς και Όλα αυτά έχουν να κάνουν, επηρεάζουν μάλλον την κοινωνία του Αφγανιστάν, όπω είπε και οι μακροοικονομικέ προβλέψει για μετά το 24. Αυτό που βλέπουμε είναι να υπάρχει έλλειψη συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσω της ε, για τη συνεργασία. Να υπενθυμίσω, Πρόεδρε, το γεγονό απλά και μόνο ότι ξέρουμε ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η αύξηση της στόχιας οφείλεται στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Είχαμε κάνει μια έρευνα με την δική μας ε, στήριξη, βέβαια, είχαν κάνει μια έρευνα με την δική μας στήριξη το 2017 γι' αυτό. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση με τις διεθνείς πολιτικές. Δηλαδή, είχαμε το πλαίσιο που θεσπίστηκε το 16 ασφάλειας και συνεργασίας με 10 εθνικά σχέδια προτεραιότητας ανατομέα και κάναμε την διάμεση αναθεώρηση με το συνδεμένο πρόγραμμα για να καθορίσουμε τις προτεραιότητες για την κυβέρνηση. Όσον αφορά την στήριξη των γυναικών στο Αφγανιστάν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μείγμα διαφόρων προσεγγίσεων και η εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας αφορά ακριβώς την οικονομική ενίσχυση των γυναικών και αυτό το εποπτεύουμε μέσω και εθνικών συμβάσεων ώστε να κάνουμε μια αξιολόγηση για αυτή την κατάσταση και έχουμε επίσης και κάποια επιμέρους μικρότερα προγράμματα τα οποία εξετάζουν και ασχολούνται με την ενίσχυση των γυναικών, τη συμμετοχή του στη δημόσια ζωή, στην κοινωνία των πολιτών κτλ. Ήδη δηλαδή είχαμε κάποιες πολύ θετικές εμπειρίες με την εφαρμογή διαφόρων συμβάσεων που δεν θα ήθελα να αναφέρω λεπτομερώς αλλά να τονίσω μόνο ότι όλα αυτά συμβαδίζουν με συγκεκριμένες τεχνικές αρρωγές και μεταρρυθμίσεις όσον αφορά διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, την ε, θέσπιση ενός οργάνου ε, ελέγχου Ελεκτικού Συνεδρίου στο Αφγανιστάν για την καταπολέμηση τη διαφθόρα. Και για τα συγκεκριμένα ερωτήματά σας, Πρόεδρε, να πω ότι τα μέλη του ΟΗΕ αυτή τη στιγμή αποτελούν το μεγαλύτερο εταίρο ανάπτυξη ε, του Αφγανιστάν. Είχαμε και διάσκεψη στο Βρυξελών το 2016. Αν λάβουμε υπόψη μας λοιπόν την συμβολή, τη συνεισφορά από τον προπολογισμό της Ένωσης, αυτό σημαίνει ότι η μεγαλύτερη εταίρη είναι η ΕΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Δεν έχω ακριβή στοιχεία, αλλά απλά και μόνο σας το λέω για μια γενική εικόνα. Ευχαρίστω να σας δώσω περαιτέρω στοιχεία αν θέλετε. Τώρα για την ειρήνη. Ελπίζουμε να έχουμε πρόοδο και Έχουμε και την διάσκεψη της Γενέβης που ανέφερε συνάδελφος. Να τονίσω μόνο ότι μπορεί να βρήκαμε κάποια λύση για την ειρήνη, αλλά θα πρέπει όλα αυτά να μεταφορθούν με τη δική μας συμβολή επίσης και στην κατάσταση της κοινωνίας και της οικονομίας. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Τζούντι, όμως πριν σου δώσω το λόγο, Πριν σου δώσω το λόγο, μήπω να δώσουμε το λόγο στην Κάριτα από την Πολωνία. Σα ευχαριστώ που ήρθατε, αλλά όχι Τζούντι, θα έχει το λόγο. Ωραία. Συγγνώμη που και συγγνώμη που θέτω ερωτήματα που μπορεί να ήδη έχουν απαντηθεί. Αν έτσι πείτε το μου και στην Επιτροπή Δημοσίων ε, Ελευθεριών αύριο θα, συνεχί... θα συζητήσουμε την κατάσταση στο Αφγανιστάν μετά από προσπάθειες δύο ετών και την κατάσταση επίσης των προσφύγων. Θυμάμαι ότι είχαμε αυτή η συμφωνία για χρηματοδότηση από την Ένωση επέκταση του αεροδρομίου της Καμπούλ, το οποίο έπρεπε να μεγαλώσει ακριβώς για να υποδεχτεί όλους τους επιστρέφοντες. Και δεν θέλω να μάθω τι γίνεται με αυτό το έργο, επειδή χρηματοδοτείται από την βοήθεια για την ανάπτυξη. Οπότε πρέπει να το μάθουμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι είχαμε άτομα που επιστρέφουν που επαναπατρίζονται από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν και οι βία επαναπατρισμένοι από το Πακιστάν. Οπότε θα πρέπει να πούμε, επειδή υπήρχε εδώ μια διευκόλυνση, μια χρηματοδότηση από την Ένωση για αυτές τις διαδικασίες, πώς εξελίσσεται η ενσωμάτωση αυτών των προσφύγων, οι επαναπατριζόμενοι λοιπόν και από την Ένωση αλλά και από τις γειτονικές χώρες, πώς εξελίσσεται η ενσωμάτωσή τους και τι γίνεται με την κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν που όχι μόνο δεν βελτιώνεται αλλά επιδεινώνεται. Οπότε να μου πείτε τι επιπτώσει έχει αυτό στους επαναπατριζόμενους. Ωραία, λέει πρόεδρος η Κομισιόν. Μήπως θέλει να απαντήσει, δεν ξέρω αν είναι καταλληλότερη. Πάντως, για τη χρηματοδότηση πρέπει να ακούσουμε λεπτομερώς τι έγινε. Δώσατε κάποια στοιχεία, αλλά πείτε μας κάτι παραπάνω, ιδιαίτερα για το αεροδρόμιο. Βεβαίως, Πρόεδρε, δεν μπορώ να προκαταβάλω συζητήσεις που θα γίνουν αύριο. Δεν έχω τέτοια εντολή βέβαια. Αλλά συνοπτικά να υπογραμμίσω ότι η βοήθεια για την ανάπτυξη κυρίως αφορά επαναπατριζόμενους και εκτοπισμένους στο εσωτερικό του Βένσταν για την μακροχρόνια ενσωμάτωσή τους. Έχουμε κάποια άλλα μέτρα που συνδέονται με αυτό, κυρίως για το Ιράν και την κατάσταση των Αυγανών που έχουν μετακινηθεί εκεί. Αν δούμε λοιπόν το πακέτο Αυτό ήταν 210 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Από το 16 έχουμε τρεις φάσεις. Άμεση ενίσχυση και ανθρωπιστική βοήθεια αμέσως μετά την άφηξη αυτό το ατόμο στο Αφγανιστάν. Υπάρχουν κάποια μέτρα με κάποιες ανάγκες που αντιμετωπίζουμε άμεσα ας πούμε, κατάρτιση, στήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων κλπ. Και μετά έχουμε την μακροχρόνια ενσωμάτωση, όπου συνεργαζόμαστε με τοπικές κοινότητες που αφορούν τους επαναπατριζόμενους. Με αυτό ανοιχτό σε όλους τους δικαιούχους, αλλά θα είδατε ότι ο κυριότερος όγκος των ατόμων που αφορούν αυτά τα μέτρα είναι τα άτομα που απαναπατρίζονται από το Πακιστάν και το Ιράν όταν επιστρέφουν δηλαδή αυτά τα άτομα στο Αφγανιστάν και να τονίσω ότι επίσης καλύπτουμε και το Ιράν και τις, ε, τα κυκλικά σχήματα, κυκλικές μορφές μετανάστευσης εκεί. Επίσης, στηρίζουμε την επέκταση του αεροδρομίου στην Καμπούλ Αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο χώρο στις αφήξεις για την στήριξη των επαναπατριζομένων για τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις κλπ. Αυτά πρώτα ευχαριστώ. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό απάντησε το ερώτημά σας. Όχι, δεν μου το απάντησε. Γιατί άκουσα τους όρους ενσωμάτωση μετά τον επαναπατρισμό. Δεν μου είπατε κάτι για τον ίδιο τον επαναπατρισμό, αλλά θέλω να μου πείτε τι γίνεται με την ενσωμάτωση. Όταν ενσωματώνονται άτομα στην κοινωνία, ε, αυτή η κοινωνία είναι όλο και λιγότερο ασφαλής. Οπότε αυτό είναι μια πρόκληση. Τι γίνεται. Ίσως στη Λίμπη θα μπορούσατε να το συζητήσετε. Ξέρω ότι είναι επίμαχο αυτό το ζήτημα. Εδώ και μισή χρόνια νομίζω είχαμε μια συζήτηση αυτό. Είχαμε και την χρηματοδότηση για τις απελάσεις και η Κομισιόν νομίζω δεν χρηματοδοτούσε πια αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά για τη χρηματοδότηση, αλλά Περίπου αυτό ίσχυε τότε. Ε, ελπίζω να, να, μην κάνω λάθος. Ναι, αλλά μου φαίνεται, Λίντα, ότι αυτό είναι μια απεικόνηση του προβλήματο που αντιμετωπίζουμε ω Κοινοβούλιο. Γιατί αύριο δεν θα μιλήσουμε για την ενσωμάτωση μέσω τη βοήθεια για την ανάπτυξη αυτών που επαναπατρίζονται στο Αφγανιστάν. Θα συζητήσουμε άλλα ζητήματα, όπω το πώ, α πούμε, επιστρέφουν από την Ένωση στο Αφγανιστάν. Αλλά κάποιο τέλο πάντων πρέπει να παρακολουθήσει ε, πώς ταπανούνται αυτά τα χρήματα για του επαναπατριζόμενου στο Αφγανιστάν και, αν κατα... και κατά πόσο του προσφέρει κάποιε νέε ευκαιρίε στη ζωή του. Ανεξάρτητα από που επαναπατρίζονται. Εντάξει, τώρα αν δεν έχουμε ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή, εντάξει, αλλά εμεί αφιερώνουμε κονδύλια εκεί και είναι κάπω δύσκολο να ενσωματώσουμε κόσμο σε κοινωνία που δεν θέλει, γιατί δεν θέλανε να επαναπατριστούν και μια κοινωνία που είναι φτωχή και γίνεται όλο και φτωχότερη. Ναι, Judith, ίσως θα πρέπει να ρωτήσεις χωριστά την Κομισιόν για αυτό το θέμα από την Επιτροπή μας. Ας θα δώσουμε χρόνο της Επιτροπής να απαντήσει της Κομισιόν. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Αν θέλετε θα έλεγα ότι ήταν συγκεκριμένο το ζήτημα. Αφορά όμως μια περίπλοκη υπόθεση και θα σας απαντήσουμε σε αυτό το χρόνο. Ωραία, θα επανέλθουμε, λέγει η Πρόεδρος. Θα πρέπει πραγματικά να ξέρουμε, έχεις δίκιο, πού πάνε τα χρήματα. Με ποια προγράμματα, ποιος τα διαχειρίζεται, πώς δαπανώνται τα κονδύλια, τι αντίκτυπο έχουν τα προγράμματα κλπ. Ωραία. Φρανκ, ο εισηγητής μας, θες να προσθέσεις κάτι. Όχι. Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι ελπίζω ότι κάποια στιγμή όλα όσα επενδύουμε εμείς, όλα όσα επενδύουν άλλοι, με δεδομένο βεβαίως ότι τα χρήματα αποστέλλονται, θα καταλήξουν στη σταθεροποίηση της προκειμένης χώρας, γιατί όσα έχουμε δει από το 2011 ε, καταδεικνύουν το αντίθετο. Είτε είναι αποφασισμένοι να έχουν μια δημοκρατικά ελεγμένη ηγεσία, είτε υπάρχουν στρατεύματα που εγκαθίσταται εκεί, είτε φεύγουν τα στρατεύματα. Η αλήθεια είναι ότι το Αφγανιστάν παραμένει εξαιρετικά ασταθές και δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει και από αυτό το καταπιστικό καθεστώς. Και κάποια στιγμή θα προκύψει το ερώτημα κατά πόσο αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε οικονομικά. Γιατί αν η στήριξή μας σημαίνει ότι κάθε φορά χρησιμοποιούμε, κινητοποιούμε δισεκατομμύρια ευρώ, ε, τότε κάποια στιγμή θα θέλουμε να δούμε αποτελέσματα. Και αν στατιστικά τα αποτελέσματα αυτό που μας δείχνουν είναι ότι τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας αυξάνουν, τα άτομα που ζουν σε ε, συνθήκες επισφάλειας αυξάνουν, ε, τότε ε, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συζητάμε ανοιχτά και είναι και ένα ζήτημα ασφάλειας, είναι ένα ζήτημα γεωγραφικής, γεωγραφικού ελέγχου. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε το λαό του Αφγανιστάν. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι πολύ αισιόδοξα. Συχνά συζητάμε και για τους Αμερικάνους και μιλάμε και για τον προπολογισμό άμυνας, αλλά όταν ε, συζητάμε για το λεγόμενο soft power και την ανθρωπιστική βοήθεια, η Ευρώπη ε, έχει αναλάβει σημαντική δράση στο Αφγανιστάν. Καλώς, συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε έτσι και με το σημείο 20. Στις 17 Οκτωβρίου στις 12 θα πρέπει να έχετε καταθέσει τις τροπολογίες σας. Το επόμενο σημείο που θα συζητήσουμε είναι μαζί με την Επιτροπή ΦΑΜ στις 21, στις, με συγχωρείτε το σημείο 21, όπου θα συζητήσουμε για την εξάλληψη της βίας ενάντια στις γυναίκες και στα νερά κορίτσια. Α, εν ώψη και της Διεθνούς ημέρας για τις νέες κοπέλες για, που είναι την ε, Πέμπτη. Η, θα, η συνεδρίασή μας θα συνεχίσει στις 4 η ώρα. Μέχρι τότε έχουμε ένα διάλειμμα. Ευχαριστώ.